ψηφίσματα τα οποία θα, θα τεθούν σε ψηφοφορία μετά από τη συζήτηση. Τώρα έχουμε τη συζήτηση για τη Βυρμανία και πρώτη είναι η κυρία Ντεκάιζερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βυρμανία συνεχώς ε, χειροτερεύει. Να σας θυμίσω την καταπίεση της βυρμανικής κυβέρνησης προς το λαό. Να σας θυμίσω τι έγινε με το βραβείο Ζαραχάροφ στην Κιμσούκη. Να σας θυμίσω ποια είναι η στάση της κυβέρνησης εν ώψη των εκλογών. Σε αυτή τη φάση η δημοκρατία ο εκδημοκρατισμός ε, θα, της ε, κυβέρνησης στην Βυρμανία θα έπρεπε να καταλήξει σε εκλογές. Και άμα αυτό όμως γίνει με ένα σύνταγμα που έχει συντάξει ο στρατός, όπως φαίνεται και να συμβαίνει, τότε τότε μη σημαίνει ότι δεχόμενοι αυτά τα πράγματα νομιμοποιούμε το στρατιωτικό καθεστώς και δίνουμε νομιμότητα στο 25% των εδρών που οι στρατιωτικοί θα πάρουν στο κοινοβούλιο. Σημαίνει ότι θα ανεχθούμε την υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, τόσο ώστε να μην έχουμε μια πολιτική φάρσα σε όλη τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι οι πρώτες εκλογές μετά από 20 χρόνια και πρέπει κανείς να είναι αισιόδοξο ότι υπάρχει μια μεταβατική κατάσταση προς, προς τη δημοκρατία. Τίποτα όμως δεν διασφαλίζει ότι οι εκλογές αυτές θα είναι δημοκρατικές και θα οδηγήσουν σε πραγματική αλλαγή. Ε, στο ψήφισμά μας έχουμε καταγγείλει πολλές περιπτώσεις παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν καθημερινά στη Βιρμανία. Ε, δεν ε, μπορούμε να, ε, να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία ο λαός της Βιρμανίας. Ποιος να τους βοηθήσει. Οι γειτονικέ χώρες και οι οποίες βοηθούν, εμπορεύονται και χρηματοδοτούν τη χώρα, αυτά, τη χώρα αυτή είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε, άρα αυτές πρέπει να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Ευχαριστώ τώρα κυρία Βεζιά για δύο λεπτά. Από το 1962 η Βρισμανία βρίσκεται υπό μία στρατιωτική χούντα, ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα του κόσμου. Όσοι δημοκράτες σήκωσαν κεφάλι, συνελήφθησαν, και 230 βουδιστές ε, καλόγεροι ε, που συμμετείχαν στις ε, ειρηνικές διαδηλώσεις του 2008 είναι ακόμα φυλακισμένοι. Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τη Βυρμανία πρόσφυγες ζουν στο Μπαγκλαντές, στη Μαλαισία σε άσχημες συνθήκες. Χιλιάδες άτομα μετακινήθηκαν χωρίς τη βούλησή τους απειλούνται δημοσιογράφοι. 14 δημοσιογράφοι τουλάχιστον βρίσκονται σήμερα στη φυλακή. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω την Λάλα Ουίνα, 25χρονη δημοσιογράφο που καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλακή για παράνομη εισαγωγή μίας μοτοσικλέτας. Και, γιατί, και αυτό γιατί τόλμησε να πάει σε ένα μοναστήρι, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. Η Χούντα έχει εξαγγείλει εκλογές όπως είπε και η κυρία Ντεκάιζερ, δεν έχουν στόχο αυτές οι εκλογές παρά να νομιμοποιήσουν το υπάρχον καθεστώς. Εμείς ε, σήμερα για μια ακόμη φορά πρέπει να καταδικάσουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βυρμανία, να καλέσουμε την κυβέρνηση σε διάλογο να σταματήσει την πολιτική των παιδιών στρατιωτών. Να καλέσουμε τη ρωσική, ειδική και κινέζικη κυβέρνηση να ασκήσουν την επιρροή τους. Αλλά κύριε Επίτροπε, εγώ σας παρακαλώ να είστε εσείς ο εκπρόσωπός μας στην Κομισιόν την ίδια και το Συμβούλιο, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα έναντι της κυβέρνησης της Βυρμανίας. διότι δεν έχουμε καμία απόδειξη, χειραπτή απόδειξη ότι γίνεται δημοκρατικός διάλογος. Ζητούμε λοιπόν να εφαρμόσετε τα πάντα ούτω ώστε και κόβετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τάνοκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, έχω χάσει πια το μέτρημα. Πόσες φορές έχουμε εδώ συζητήσει σε αυτό το οίκο την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βυρμανία. Να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε κάνει εμείς για να θυμόμαστε πάντοτε γιατί πρέπει να πιέζουμε συνεχώς τους στρατηγούς. Αναφέρομαι στην Aung San Suu Kyi, της οποίας η φωτογραφία έχει αναρτηθεί και εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, ηγέτης της αντιπολίτευσης, η οποία έχει υποστεί τόσες διώξεις. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε εξ ονόματος αυτών. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για μειονότητα των Ροχιγκίγια που ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων, που διώκονται από, το στρατό. Πολλοί είναι διεσπαρμένοι στο νοτιοανατολικό Μπαγκλαντές. Ως δημοκράτες καθήκον μας είναι να καταδικάζουμε τέτοιου είδους πράξεις παντού στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Επόμενος θα μιλήσει ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα για δύο λεπτά. Πριν από μερικού μήνε επισκέφθηκα στα σύνορα μεταξύ Ταϊλανδία και Βυρμανία μερικού από του χιλιάδε πρόσφυγε που περιμένουν ακόμα να γυρίσουν στα σπίτια του. Ή απλώ περιμένουν να επιβιώσουν μια μέρα παραπάνω. Συναντήθηκα με μερικές από τις αντιπολιτευτικές οργανώσεις, τον Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία για παράδειγμα, ε, της οποίας μέλος είναι και το βραβείο Ζαχάροφ. Και εγώ λέω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με ιδιαίτερη σοφροσύνη, να μην υποστηρίξουμε εκλογές που οργανώνει η ίδια η Χούντα και με όρους αν και αυτούς που σήμερα παραβιάζουν τους βασικούς όρους της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συναθρίζεσθε. Αποτελούν λοιπόν κίνδυνο όλα αυτά για οποιαδήποτε δημοκρατική μεταρρύθμιση της χώρας. Πράγματι έγιναν κάποιες μικροαλλαγές. Το 2009 ε, απελευθέρωσαν ε, καμιά εκατοστή κρατουμένους ελάχιστοι από αυτούς ήταν πολιτικοί κρατούμενοι βέβαια σήμερα έχουμε γύρω στις 2.000-2.100 ε, πολιτικούς κρατούμενους και κρατούμενες στη Βυρμανία είναι αδύνατο λοιπόν εμείς να θεωρήσουμε σωστές, ελεύθερες και δημοκρατικές αυτές εκλογές. Πρέπει να θυμίσουμε ότι το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για να γίνουν αυτές οι εκλογές. Οποιοδήποτε διάλογος να προχωρήσουμε στην κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος, αλλά όμως με την ανεφόρον πολευθέρωση αυτών των πολιτικών κρατουμένων και τη δυνατότητα των προσφύγων να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και λέω στην Κομισιόν, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η μείωση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση αυτών των προσφύγων. Είναι κατεπίγουσα η κατάσταση. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που απαιτούν τη συνεργασία μας. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην ε, περιορίσουμε αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, καταρχήν ο κύριος Μάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βερμανία έχει επιδεινωθεί δραματικά. Η πολιτική καταστολή με σερβιτική και σεξουαλική βία, ε, παιδιά τα οποία ε, γίνονται στρατιώτες, 2.000 ε, πολιτικοί κρατούμενοι. Οι πρώτες ελεύθερες εκλογές το φθινόπωρο αυτού του χρόνου είναι πραγματικά αστείο. Επίσης είναι η κατάσταση των όσων ε, μένουν στο, σε στρατόπεδα προσφύγων. Πολλοί πηγαίνουν στο Μπαγκλαντές όπου διώκονται βάναυσα. Χαιρετίζω την προθυμότητα της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές να υποδεχτεί την δική μας αντιπροσωπεία για εξέταση της κατάστασης. Αύριο θα πάμε στο Ντακάρ για να μεταβούμε στο Κόξ Μπαζάρ και στην περιοχή Μπανταμπάρ για να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι. Ωστόσο είναι σαφές ότι οι διοκόμενοι χρειάζονται διεθνή προστασία προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συνεπής όσον αφορά την απόρριψη των αρχών της Βερμανίας έως ότου γίνουν ορατοί, ορατές προόδοι στην υπόθεση της δημοκρατία. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παλέτσκης. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε. Ναι, όπως ε, και όλοι οι συνάδελφοι θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που δυστυχώς ε, σε αυτή την ώρα είναι σχεδόν άδεια ε, συζητούμε κατ' επανάληψη στην ε, τρομακτική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία. Εγώ ίδιος πρόσφατα μίλησα σχετικά αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι μετά από αυτή τη σημερινή συζήτηση η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος. Γιατί, γιατί για πρώτη φορά ε, συζητούμε για τόσο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας παράλληλα τη συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλεία, την Κάθριν Άσταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αποτελεσματικότερα ε, μέσα ε, στη διάθεσή της για να βελτιώσει την κατάσταση χωρών όπως η Βερμανία παραπέζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι πεπισμένη ότι στη Βερμανία θα συμβούν ε, βελτιώσεις μόνο εάν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με μεγάλες χώρες όπως είναι η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα κλπ. Ο κύριος Πορέμπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι κλήσεις για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βυρμανία έχουν κάποια αποτελέσματα. Ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φυλακισμένοι βασανισμοί και συνεχείς ε, συλλήψεις των αντιφρονούντων. Γνωρίζουμε την κατάσταση της Αγκ Σουκί, η οποία κρατείται κατοίκων. Ε, και στην οποία απεγκάλυφθηκε κατηγορία ε, απόφαση φυλάξης τριών ετών. Επίσης, οι εθνωτικές μειονότητες διώκονται συστηματικά. Εκείνοι που έχουν ε, χριστιανικές πεπιθήσεις επίσης διώκονται και πάρα πολλοί προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στην Ταϊλάνδη. Οι αρχές της Ταϊλάνδης θέλουν όμως να απελάσουν τους ε, Καρέμ ε, Κάρεν ε, και νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο οφείλουμε να μεριμνούμε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε τον κύριο Κορχόλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε σοβαρέ ανησυχίε όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία. Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Ε, έχουμε απλώς ε, φωτίσει ορισμένα θέματα, αλλά νομίζω ότι ο πιο σημαντικός σκοπός αυτού του ψηφίσματος είναι να αποστείλει ένα χειρό μήνυμα ότι πραγματικά ανησυχούμε για την κατάσταση στη χώρα αυτή. Επίσης, ε, ανησυχούμε για την απόρριψη του θέματος να επαναπατριστούν οι πρόσφυγες στη Βερμανία. Οι πρόσφυγες Καρέν ε, απειλούνται από καταναγκαστική εργασία και ε, ίσως ε, και, και, ενδεχομένως θα αναγκάζονται να πάνε στο στρατό. Νομίζω ότι, είναι, ότι ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παράσουμε μια βοήθεια και στις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο κύριος Ταραμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά η Βιερμανία είναι στο κέντρο της προσοχής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο στα κατεπήγοντα και για μια ακόμη φορά εκφραζόμαστε κι εμείς για τη Βυρμανία, για το πώς μεταχειρίζεται τους πολίτες της κλπ. Εκεί όπου χώρες εξελίσσονται με το χρόνο, η Βερμανία τίποτα. Η νικήτρια του βραβείου Ζαχάροφ είναι κατοίκου σε κατοίκον περιορισμό, πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πολιτικοί κρατούμενοι, έχουμε τα παιδιά στρατιώτες και χίλιες δυο παραβιάσεις που δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ. Εμείς θέλουμε οι επόμενες εκλογές να γίνουν ελεύθερα, να υπάρχει εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, θα πρέπει οι παρατηρητές να διαπιστώσουν ότι οι εκλογές είναι ελεύθερες και όχι νοθευμένες. Ούτως ώστε να μην νομιμοποιήσουμε μέσα από την κάλπη το καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφη. Ε, συνάδελφε, επόμενη, μιλήτρια η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό. Η στρατιωτική χούντα έχει κυβερνήσει τη χώρα αυτή με τη βία και την οθεία. Εγώ ζητώ γενικές και ελεύθερες κοινοβουλευτικές εκλογές για το 2010 έτσι ώστε να υπάρξει μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση στη Βυρμανία. 27% του Κοινοβουλίου είναι μέλη του στρατού, προέρχονται από το στρατό, είναι άμεσες επιλογές της ε, κυβέρνησης και μας δίνουν μια σαφή ιδέα για το πόσο νομιμοποιημένη είναι η κυβέρνηση αυτή. Δεύτερον, ε, γνωρίζω ότι η στρατιωτική χούντα ε, της ε, χώρας αυτής το 2005 υπέγραψε την συνθήκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών, όμως δεν την επικύρωσε. Η διαφθορά θα πρέπει οπωσδήποτε να χτυπηθεί, γιατί είναι η ρίζα πολλών κακών. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Γκέριγκερ για ένα λεπτό. Μετά από 20 χρόνια γίνονται ελεύθερες εκλογές και αυτό είναι ένα βήμα για τον εκδημοκρατισμό. Φτάνει όμως αυτές οι εκλογές να είναι ανώθευτες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και οι Σανσούρκη και όλοι και όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που βρίσκονται στη φυλακή. Κατά δεύτερο, οι εκλογές ε, θα πρέπει να είναι ανοιχτές ε, και στους ε, πρόσφυγες Βυρμανούς που έφυγαν λόγω βασανιστήριων σε άλλες χώρες όπως τον Μπαγκλαντές. Ε, επίσης ο στρατός δεν θα πρέπει να έχει εγγυημένο το 25% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί η είσοδος στους διεθνείς παρατηρητές. Θέλουμε λοιπόν ελεύθερες εκλογές στη Βυρμανία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Τώρα έχουμε τον κύριο Σόγκορ στο πλαίσιο του Catch the Eye. 2010 folyamán szabad, demokratikus választásokat η στρατιωτική χούντα μας υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές το 2010. Είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση ούτως ώστε να υπάρξει πράγματι δημοκρατική μετάβαση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι θρησκευτικέ και εθνοτικές μειονότητες να έχουν δυνατότητα να λάβουν μέρος ε, στις εκλογές. Αυτό θα βάλει ένα τέλος στις εθνικές ε, σειράξεις. Έχουμε κυνηγιστικές μειονότητε. και νομίζω ότι η Κίνα θα μπορούσε επίση να παράσχει μια βοήθεια και είναι σημαντικό, ωστόσο, και η ίδια η Κίνα να αναγνωρίσει τις τις μειονότητες του Σουγκούρ και την, του Στιβατανούς. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ασκήσει μια πίεση που θα είναι πιο αποτελεσματική, εφόσον σέβεται και στη δική της επικράτεια ε, τις δικές της μειονότητες. Γιατί υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι νόμοι για, που επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένες μειονοτικές γλώσσες ε, ε, και σε ορισμένα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ορισμένες μειονότητες δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλούν τη δική τους γλώσσα και στο βαθμό αυτό δεν μπορεί να διατηρήσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, η στρατιωτική χούντα στη Βερμανία οδήγησε στη πραγματική επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν διώξεις ε, θρησκευτικών μειονοτήτων, ε, γίνεται εθνοκάθαρση, ε, χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι βασανίζονται ή κρατούνται παράνομα. Όλα αυτά ανήκουν στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα πρόκειται να διεξαχθούν κάποιες φαινομενικά νόμιμες εκλογές που δεν πρόκειται όμως να βελτιώσουν την κατάσταση Νομίζω ότι τέτοιου είδου ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να χρησιμεύσουν. Θα πρέπει να επιδείξουμε μια πραγματική πολιτική βούληση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να επηρεάσουμε την Ινδία αλλά και την Κίνα για να μπορέσουν να πιέσουν την κυβέρνηση της Βυρμανίας προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά και οι μεθοριακές χώρες της Βυρμανίας θα πρέπει να πιεστούν ούτως ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ε, τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Φρέντερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγο καιρό κάποιοι είπαν ε, ότι ξαναήχαμε ψήφισμα για τη Βερμανία. Αλλά διαρκώς θα πρέπει να μιλάμε για τη Βερμανία, γιατί είναι μία από τις χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη καταστολή. Είναι μία από τις χώρες όπου συστηματικά παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για χαρακτηριστικά της καθημερινότητας της Βυρμανίας, ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταχρηστικές ε, ε, συλλήψεις, εξοδικαστικές συλλήψεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι τα μέλη της βουδιστικής κοινότητας διώκονται συστηματικά. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ε, η σωστή διεθνής παρατήρηση έτσι ώστε να γίνουν σωστές ε, εκλογές. Διαφορετικά αυτή η στρατιωτική κούντα θα παραμείνει στην εξουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ρέντινγκ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, όπως τόνισαν τα ε, μέλη εδώ, οι βουλευτέ εδώ, υπάρχουν σοβαρέ παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζουν στη Βερμανία. Η στρατιωτική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στις διεθνείς εκκλήσεις να τεθεί ένα πέρα σε αυτές τις παραβιάσεις και δεν απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατούμενους, ε, ακόμα και την Ουγ Κι. Ε, Επίσης η μειονότητα των ε, Κάρεν ε, πιέστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συνεχίζει. 80% του πληθυσμού ζουν ε, στην Ήπεθρο και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά επανάληψη έχει εκδώσει κάποια ψηφίσματα που καταδικάζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης ε, έχει ασκήσει κάποιες κυρώσεις και έχουμε ασκήσει πίεση σε άλλες χώρες μεθοριακές της Βερμανίας όπως είναι η Ινδία και η Κίνα να ασκήσουν πίεση επίσης. Κάτι που πράττουν πράγματι ορισμένες από αυτές τις χώρες. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα μέτρα έχουν δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες για τη στρατηγική κυβέρνηση αλλά δεν ε, μπόρεσαν να επιφέρουν ριζικές μεταβολές. Τώρα, η στρατηγική κυβέρνηση υποσχέθηκε τη διεξογή εκλογών εντός του 2010 σαν ένα βήμα προς ε, μια βαθμιαία μετάβαση προς τη δημοκρατία. Ε, δεν μπορούμε παρά να ασκήσουμε μια κριτική σε αυτές τις εκλογές όταν όμως ε, δημοσιευθεί ε, ο, δημοσιοποιηθεί ο νέος εκλογικός νόμος. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με την ε, κυβέρνηση προκειμένου να τυπήσει, να αξιοποιήσει την ευκαιρία των εκλογών για να αλλάξει την κατάσταση αυτή και να γυρίσει μια θετική σελίδα στην ιστορία της Βερμανίας. Λέγοντας το αυτό, θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να απομονώσει τη Βερμανία και είμαστε πράγματι οι μεγαλύτεροι δωρητές ανθρωπιστικής ε, συνδρομής, αρρωγής προς αυτή τη χώρα. Το, ο μεγαλύτερος όγκος της ε, βοήθειας αυτής πηγαίνει στην Ήπεθρο ε, κυρίως στα, στις περιοχές του Δέλτα που επλήγησαν από τον ε, τυφώνα, αλλά και στις συμμεθοριακές περιοχές όπου είναι εγκαταστημένοι πάρα πολλοί πρόσφυγες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η έκθεση του ειδικού εισηγητού των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται, ε, ομιλεί μια πολύ ξεκάθαρη γλώσσα και υποστηρίζουμε την έκθεση του ειδικού εισηγητού των Ηνωμένων Εθνών και είμαστε πρόθυμοι να τον συνδράμουμε στο έργο του. Αλλά γνωρίζουμε ότι άμεσε δραστηριότητε στα επίπεδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία ε, δεν είναι δυνατέ. Για παράδειγμα, δεν θα προσκληθούμε ως παρατηρητές στις εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε έμεσα μέσα. Γι' αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, συμπεριλαμβάνονται ε, ως όρος ε, σε όλα τα προγράμματα παροχής βοήθειας, ώστε να προωθήσουμε το διάλογο και τις δημοκρατικές αξίες. Για να το κάνουμε πρέπει να αποστείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και το Κοινοβούλιο, το οποίο φάνηκε, εμφανίστηκε ενωμένο σήμερα, έχει ένα τέτοιο ξεκάθαρο μήνυμα και με βέβαιο ότι θα εισακουστεί. Επίσης είμαι βέβαιο ότι δεν θα πρέπει να εκχωρήσουμε σε άλλους ε, το δικό μας ε, καθήκον ε, προς άλλες χώρες. Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δεσμευτούμε άμεσα όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε και ε, ε, κατατάθηκαν έξι ψηφίσματα, η συζήτηση περατώθηκε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στη συνέχεια. Ακολουθεί η ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα για την Βενεζουέλα. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Ε, υπάρχει κοινό ψήφισμα τριών πολιτικών